κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, 55 ξανά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 62 σε δύο ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 62. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. είναι δεύτερο τμήμα στην παράγραφο 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη εν. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Z υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΒ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΕΦ, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη AH υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράθεμα 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για όλο το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κυρία Σαπόσκα. Σε le Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω πως ε, καταθέτω αυτή τη στιγμή και γραπτά την άποψη της μειοψηφίας. We take note that and of course allowed to do that. Βεβαίως και έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι Σαουδική Αραβία και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ρόλο στη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. κυρία Ματέρα είναι εδώ. Sorry. On, on where? To replace Amendment 10. Here. Okay. Yeah, Mrs. Par Mrs. Parvanova. Κυρία Πάρνοβα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ε, ξεχωριστά τα 16, 17 και 18 στην συμβιβαστική 4, γιατί εδώ ο τρόπος με το οποίο έχουν συμπεριληφθεί δεν μας καλύπτει. Λυπάμαι πολύ, αν μπορείτε λοιπόν αυτά να τα ε, ψηφίσουμε ξεχωριστά. Δηλαδή δεν υπάρχει συμβιβαστική τροπολογία, θέλετε χωριστή ψηφοφορία για τα 16, 17 και 18. Καλά σας κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία. Ξεκινάμε. Ε, συμβιβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 10. Εκεί έχουμε μια προφορική της κυρίας Κιλ Νίλσεν. Σας ρωτώ καταρχήν, συμφωνείτε να υποβάλουμε την προφορική? Ωραία. Άρα λοιπόν την 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και μετά πηγαίνουμε όπως ζητήσατε και εσείς 16, 17 και 18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 κατά αποχές εγκρίνεται 31 λοιπόν. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ την 31 την κάναμε ωραία 32 λοιπόν 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασική 1 υπέρ 2 κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα για όλο το ψήφισμα θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει. Έληξε. και προφανώς εγκρίνεται. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο που είναι η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Παπαδοπούλου. Όχι. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν κατευθείαν με την ψηφοφορία. Στην 6. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρώτη επέρ, κατά, αποχές. Ξεχάσαμε, ξεχάσαμε την 7. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα λοιπόν περνάμε τώρα στην συμβιβαστική 2, λέει ο Πρόεδρος. Είναι προφορική για την 9 έχουμε. Υπάρχουμε για την τροπολογία 9 προφορική. Μπορούμε. Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε και την προφορική τροπολογία του 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην τροπολογία 16 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21, εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ, τμήματική λοιπόν, κατά, εγκρίνεται. Η δεύτερη υπέρ, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 22, τροπολογία 22 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 23 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 24, 25 τροπολογία υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 και εδώ έχουμε τμηματική για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η δύο υπέρ κατά αποχές υπέρ εγκρίνεται, Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα λοιπόν για όλο το ψήφισμα ανοίγει η ψηφοφορία. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Περνάμε στο ε, επόμενο που είναι για την ε, δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία κτλ. Η κυρία Κέκους είναι η συντάκτρια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε απευθείας με την ψηφοφορία. Η τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Εδώ για την 32 θέλω ηλεκτρονικά, παρακαλώ, 32 ηλεκτρονικά. Έκλεισε. Απορρίπτεται. 33. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34. Είναι προφορική. Έχουμε αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζεται η 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά για 34. Ξεκινάμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Λυπάμαι. Περνάμε στην τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά. Για την 36. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 36. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά για την 39. Παρακαλώ ξεκινάμε την ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται.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 Ψηφίζουμε λοιπόν τη 46 υπέρ. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα λοιπόν τμήματικά τη 47, ένα τμήμα μόνο. Για εκείνο το τμήμα του 47 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το κομμάτι αυτό. Το 15 καταπίτη ή 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 καταπίπτει 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 είναι και εδώ χωριστή η ψηφοφορία υπέρ για το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται και για το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 καταπίπτει 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 24 υπέρ κατά αποχές Νομίζω για την τροπολογία 24 ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει για την 24. Κλείνει. Amendment 2 in favor. Λοιπόν, στην επόμενη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ακόμα. Λοιπόν, για την 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25. Καταπίπτει. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 καταπίπτει. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 5 καταπίπτει, η 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 6 καταπίπτει, η 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 29 ήταν και για ένα τμηματικό, πηγαίνουμε στην 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 καταπίπτει οπότε για όλο το ψήφισμα ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία ξεκινάει κλείνει εγκρίνεται <coughs> Περνάμε λοιπόν στην τελευταία ψηφοφορία που είναι για την κοινωνική προστασία για όλους περιλαμβάνει και των αυτών αποσχολούμενων. Δεν βλέπω την κυρία ε, Κορνίλσεν. Να τις δώσω λοιπόν, να, σας δώσω, να ξεκινήσουμε με την ε, η πρώτη συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για να το δούμε και ηλεκτρονικά. Uh, λοιπόν, συμβιβαστική νούμερο 1. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Κλείνει. Άρα λοιπόν εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάντως που μου επιτρέπετε να ελέγχω κάθε τόσο. Περνάμε στην 12. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται, η 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, κατεβαίνουμε λοιπόν στην 19 υπέρ, τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές και εδώ τροπολογία 19 νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 19η τροπολογία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Λοιπόν, για την 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 εντάξει. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά απορρίπτεται η συμβαστική 3 θα πρέπει να ελεγχθεί ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία για την συμβιβαστική 3 κλείνει Απορρίπτεται. Το έβλεπα κι εγώ. Περνάμε στη συμβιβαστική... Στην... Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ωραία. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Για την 28 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά παρακαλώ και την 29. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 29. Λίγη. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 καταπίπτει. 32 ε, με συγχωρείτε <laughs> καταπίπτει. Λάθος μου. Γιατί 31 πρέπει να ψηφίσουμε. Είστε υπέρ της τροπολογίας 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για την 31 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Α. Την 32 παρακαλώ. Ανοίγει η ψηφοφορία. Έκλεισε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε. Λοιπόν, για την 4. Ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην συμβαστική 5 υπέρ. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιατί 5 ηλεκτρονικά. Συμβιβαστική 5. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω έχουμε την ίδια πλειοψηφία εδώ. Κλείνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 5. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη συμβαστική 6. Υπέρ στη συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε τις 48 και 6 να τις δούμε όλες μαζί. Όχι. Για τις 48 να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρώτη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η δεύτερη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο λοιπόν του ψηφίσματος ανοίγει η ψηφοφορία And the vote is closed. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους τους εισηγητές. Όλες οι εισηγήσεις σας, οι εκθέσεις σας, με συγχωρείτε, εγκρίθηκαν. Ευχαριστώ. Yeah, we're start now. Αρχίζουμε συνάδελφοι. Αρχίζουμε ξανά. Καθίστε παρακαλώ. Και αν θέλετε να συνεχίσετε να μιλάτε, έχετε όλο το ελεύθερο να το κάνετε έξω από την αίθουσα. Θα γυρίσω τώρα στα σουηδικά. Επαναλαμβάνεται λοιπόν η συνεδρίαση. Θα ήθελα να, να επιστρέψω στο σημείο 3. Στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης υπάρχει ένα αίτημα να αλλάξει η σειρά της ημερήσιας διάταξης και υποθέτω πως μπορούμε να το εγκρίνουμε. Τώρα, ε, ανακοινώσεις του Προέδρου. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε διερμηνία από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ουγγρικά, πολωνικά και σλοβακικά. Να σας πω επίσης ότι ίσως έχετε δει ένα φυλάδιο για τις γυναίκες ε, στο Ευρωκοινοβούλιο και το Παγκόσμιο Φόρουμ. Έχουν σταλεί προσκλήσεις. Το πρόγραμμα φαίνεται εκπληκτικό πραγματικά. Η εκδήλωση διεξάγεται στις 29 Νοεμβρίου και θα ήταν καλό να βρεθείτε εκεί όσοι μπορείτε, όσο περισσότερο μπορείτε. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον φόρουμ, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Νομίζω ότι θα έχει 650 συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των τριών μερών του φόρουμ. Στις 26 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τα 120 χρόνια από τότε που η Νέα Ζηλανδία έδωσε το δικαίωμα της ψήφου στις γυναίκες και η Επιτροπή μας με την, επίσης, η Επιτροπή μας με την Επιτροπή Ελίας θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί, αύριο. Και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Τώρα, όσον αφορά τις ε, αποφάσεις των συντονιστών, σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Αυτές θα σας αποσταλούν μέσω email, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Επίσης, να σας πω ότι η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τα πρακτικά της 8 Σεπτεμβρίου 2013 της 20... 2013 της 20ης και 21ης Ιουνίου 2012, 30ης Μαΐου 2012 και 23 η και 24 η Απριλίου 2012. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν, τα πρακτικά εγκρίνονται. Προχωράμε τώρα στο σημείο 12 της ημέρησης διάταξης, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Παρβανόβα, την εισηγήτρια, η οποία έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μπορώ να ζητήσω πρώτα να παρουσιάσουμε την ε, μελέτη και μετά να παρουσιάσω την έκθεσή μου. Συγγνώμη, ναι, ναι, και άρα με ενημέρωσε ήδη. Δικό μου το λάθος. Το πρώτο μέρος ήταν έτσι γεμάτο, φορτισμένο συναισθηματικά. Μάλιστα. Δεν θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα. Θα κάνω αυτό που μου είπε η Κιάρα. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Τάν από για την ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αν θυμάμαι καλά, θα παρουσιάσετε και οι δύο, πέντε λεπτά έκαστο, σε την μελέτη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ξανά εδώ εκ μέρους της Εμονάδας Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Έχω ήδη μιλήσει στο παρελθόν σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Όπως σα είπα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενική διεύθυνση η οποία θα στηρίζει τι ε, εκθέσεις ε, του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, ε, παρήχαμε μια αξιολόγηση στην έκθεση της ε, κυρίας Παρβάνοβα. Συλλέξαμε στοιχεία από διάφορες πηγές και τα συγκεντρώσαμε. Καταλήξαμε λοιπόν στο να στηρίζουμε την ε, πρόταση νομοθετική πρωτοβουλία της κυρίας Παρβάνοβα. Θα, πριν δώσω το λόγο στον ε, εμπειρογνώμονα, τον συναδελφό μου, θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τη μελέτη μας. Και είναι πραγματικά εξαιρετική χρονική στιγμή, διότι και χθε γιορτάζαμε τη μεραβία κατά των γυναικών. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι επίκαιρο. Αρχίσαμε να δουλεύουμε τη μελέτη αυτή αρκετό καιρό πριν. Συνεργαστήκαμε με την εισηγήτρια όσον αφορά την προσέγγιση και τη μεθοδολογία. Καταρχάς προσπαθήσαμε να δούμε την έκταση του προβλήματος και μετά το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη γι' αυτό και αν μπορεί να κάνει κάτι η Ευρώπη ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία του. Γι' αυτό ζητήσαμε τη συμβολή εμπειρογνωμόνων. Είχαμε τη συνεισφορά του καθηγητή Βίλμπι από το Πανεπιστήμιο του Λάνκασερ και τον κύριο Μόσερ Επίσης, ε, συλλέξαμε πληροφορίες από τα τμήματα πολιτικής που είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν, καθώς και από τις ε, νομικές υπηρεσίες, διότι η νομική πτυχή της έκθεσης είναι και η πιο περίπλοκη. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα πραγματικό και παρκτό σοβαρό πρόβλημα με πολύ μεγάλη έκταση 20 έως 25% των γυναικών έχει αποδειχθεί ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας. Και με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα υπήρξαν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή η βία και αυτά τα φαινόμενα έχουν ενταθεί από την οικονομική κρίση παρατηρείται περισσότερη ενδοοικογενειακή βία, περισσότερες, ε, περισσότερα κρούσματα διακίνησης γυναικών και αυτό φυσικά έχει και ένα σημαντικό κόστος για την κοινωνία. Τώρα, δεν μπορούμε να επιχειρηματολογούμε μόνο ε, βασισμένοι σε οικονομικά και οικονομικούς παράγοντες, οικονομικά κριτήρια. Υπάρχει και ο ηθικός παράγοντας και εμείς έχουμε προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσουμε τους παράγοντες αυτούς. Κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και πάντα προσπαθούμε να δίνουμε ακριβή στοιχεία. Όμως, εκτιμούμε ότι, περί, ότι το κόστος που επιβαρύνει τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αστυνόμευση, την ποινική δικαιοσύνη, τις κοινωνικές υπηρεσίες, ανέρχεται περίπου στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ και υπάρχει μια περαιτέρω ζημία άλλων 24 δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτό είναι το καθαρά οικονομικό κόστος της ε, έμφυλης βίας. Και αν συνεκτιμήσουμε και το ηθικό κόστος, το ποσό αυτό θα ανέβει κατά πολύ. Στο 1,8% του ΑΕΠ και πιστεύω πως ε, αυτές οι διαστάσεις και αυτό το μέγεθος φαίνεται και σε άλλες μελέτες και σε άλλους ε, τομείς. Και είναι να σας πω και μια συντηρητική εκτίμηση του κόστους της έμφυλης ευβίας. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη-μέλη δεν προσφέρουν ίσα επίπεδα προστασίας. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρος ε, ο κρατικός μηχανισμός για την εμφυλιβία. Τα νοσοκομεία έχουν δημιουργήσει ειδικά τμήματα, υπάρχουν ε, ειδικά τμήματα στα δικαστήρια, εισαγγελείς που ασχολούνται μόνο με αυτά, ενώ σε άλλα κρατημέλη, όπως οι κάτω χώρες για παράδειγμα, ισχύουν οι συνήθεις ε, ποινικέ διατάξεις χωρίς να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση που παρατηρείται σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντική η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία όμως δεν έχει την άμεση επίδραση που θα είχε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, πέραν από τα ποσοτικά στοιχεία, υπάρχουν και ποιοτικά στοιχεία, η διασφάλιση της καλύτερης προστασίας των γυναικών, και αυτό θα γίνει μέσω της ενίσχυσης του τομέα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, καθώς και της εσωτερικής και εξωτερικής συνοχής των ευρωπαϊκών δράσεων. Τέλος, όσον αφορά το τι δράσεις θα χρειαστούν. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη συμβολή τη νομική υπηρεσία και εδώ υπάρχει και η πρόταση τη εισηγήτρια ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια νομική βάση η οποία θα στηριχθεί από τις δράσεις των κρατών μελών στο τομέα της πρόληψης βίας και θα συνδυαστεί με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη βία, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιοι που θα χαράξουν τη μελλοντική πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα βοηθήσουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσχώρηση στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αυτά εν ολίγης, κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα ζητήσω από τον εμπειρογνωμονά μου, τον κύριο Μόσερ, να μας συμπληρώσει και να επεκταθεί. Σας ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και στο όνομα των συναδέλφων που με βοήθησαν να συντάξουμε την έκθεση αυτή ε, και μάλιστα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκθέσουμε τα επιχειρήματα ε, υπέρ της χρησιμότητας ενός τέτοιου ε, μιας τέτοια προσπάθεια. Βασικά αυτό θα ενίσχυε την πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ήταν ένα εργαλείο ώστε να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήταν αυτό το μέσο ακόμα ένα βήμα κατά τη γνώμη μας και εδώ αναφέρουμε και τις λεπτομέρειες. Θέλαμε επίσης να τονίσουμε που έχει να κάνει με την ε, συμβολική ισχύ του δικαίου. Αρχίζεις δηλαδή να ονοματίζεις διάφορες ζημιές που γίνονται ε, ή ε, εις των γυναικών σε διάφορες κράτη, σε διάφορα κρατημέλη και έτσι αυξάνεται και η ισότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή η βία αυτού του τύπου δεν θεωρείται ω θέμα ισότητα ή μη διακρίσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα λοιπόν, γιατί στην ουσία αυτό μετά, ε, ε, εφόσον υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κεντρικό μέσο, μετά αυτό ε, διαχέεται και στις εθνικές νομοθεσίες. Εξάλλου η ευρωπαϊκή δράση κατά αυτόν τον τρόπο θα καταστεί πιο συνεκτική, ανάμεσα δηλαδή στις εσωτερικές και τις εξωτερικές δράσεις, γιατί υπάρχουν δράσεις όπου η Ένωση παρεμβαίνει υπέρ του αγώνα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και έτσι η εξωτερική δράση θα γίνει πιο συνεπής, πιο συνεκτική με την εσωτερική. Ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φανεί πιο συνεπής όσον αφορά την ολοκλήρωση, τη δημιουργία ενός χώρου ε, όπου βαθαίνει την ελευθερία, την ασφάλεια και την δικαιοσύνη μέσω, μέσω δράσεων που σχετίζονται δράσεις για την δικαιοσύνη ε, υπέρ των γυναικών που έχουν υποστεί βία αλλά και ε, δράσεις υπέρ των δύο φύλων. Είναι επιχειρήματα αυτά λοιπόν αλλά τονίζουμε επίσης στη μελέτη μας το κόστος της αδράνειας. Ε, πολιτικά είναι επίσης μια απόφαση, μια πιθανή απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως δεν είναι απλώς μια παράληψη, αλλά μια απόφαση να μην κάνουμε τίποτα. Είναι η κατεξοχήν πολιτική απόφαση αυτή και πρέπει να το τονίσουμε κατά τη Στο δεύτερο τμήμα προσπαθούμε να δείξουμε τις ε, δυνατότητες εναρμόνισης. Ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο νομοθετικό επίπεδο για την βία κατά των γυναικών και τον ε, καταπολέμησή της, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων, οι οποίες είναι είτε τυφλές στο φύλλο, είτε αναγνωρίζουν κάποια μέρη της βίας, κάποια, κάποιες εκφάνσεις της βίας. Και η, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα πρώτο μέσο διεθνούς επίπεδου για την κατεπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το πρόβλημα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά μέσα είναι ότι ένα ευρωπαϊκό μέσο δίνει δυνατότητα της δικαστικής προσφυγής, ενώ η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης όχι. Γίνονται αναφορές ε, κρατικές, αλλά δεν δίνεται το δικαίωμα σε ένα άτομο να μπορέσει να προσφύγει με βάση αυτή τη σύμβαση στην δικαιοσύνη. Το τελευταίο μου, η τελευταία μου παρατήρηση που είναι και πιο δύσκολη ίσως είναι η δυνατότητα, η σκοπιμότητα ενός τέτοιου μέσου. Καμιά από τις λύσεις ε, των πιθανών άρθρων 82, 83 ή 90 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε το άρθρο 84 δεν δίνει πλήρη, πλήρες σύνολο αρμοδιοτήτων. Αλλά αν συνδυαστούν έτσι όπως προτείνει η συγγήτρια στην πρότασή της, φαίνεται να είναι αυτός ένα ευφιέστατος τρόπος. Αν δει κανεί άρθρα, το άρθρο 84 για την εισαγωγή κάποιων προληπτικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις να είναι καταρτισμένες, οι δικαστικές ε, αρχές επίσης, όταν τα θύματα ε, προ προβαίνουν σε καταγγελία να μην φοβούνται και οι αρχές να γνωρίζουν τα θέματα της βίας. Το, έπειτα το άρθρο 83 ομόφωνη δράση για τις σχετικές αποφάσεις και επίσης συμπεριλαμβάνονται οι τομείς της βίας που εκπορεύεται ε, από το φύλλο του ατόμου. Πιστεύουμε λοιπόν πως εν γέννη ε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έχει υποβληθεί εδώ και ελπίζουμε πως η μελέτη μας βοήθησε στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας και εκτιμούμε όλος ιδιαίτερος την εργασία που κάνετε εδώ. Προσπαθείτε να μας βοηθήσετε σε όλη αυτή την πορεία, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για την Επιτροπή μας. Θέλουμε να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση και έχουμε έρθει σε επαφή με την Κομισιόν Πολάκης με την ιδέα ότι... Ξέρετε, υπάρχουν ένα σωρό που τα καλύπτουν όλα αυτά και θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική εδώ. Τώρα, για να ξανάρθω στην αρχή, εκεί που ξεκίνησα, θα δώσω το λόγο στην κυρία Παρπανόβα τώρα. Τώρα έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, το λόμπι των Ευρωπαίων Γυναικών και και την Κομισιόν για την αξιολόγηση και τη συμβολή σε αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα για τη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όσον αφορά τις αξίες τις οποίες βασίζεται η Ένωση και το κόστος της βίας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η βία κατά των γυναικών είναι σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή έμφυλης, ε, έμφυλων διακρίσεων. Είναι ένα εμπόδιο στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. Οι γυναίκες που υπόκειται βία έχουν μακροπρόθεσμες σοβαρέ ε, σωματικές και ψυχολογικές βλάβες. Ε, επιβάλλεται έτσι κόστος ε, στις ε, αρχές υγείας, απώλεια παραγωγικότητας και μισθών. Θα ήθελα να τονίσω κάποια νούμερα εδώ. Αν και ήδη είχαμε ε, εκτίμηση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και πάλι ότι γύρω στο 20 με το 25% των γυναικών στην γυναίκα έχουν ε, πέσει θύματα σωματικής βίας και 10% έχουν υποστεί σεξουαλική βία με άσκηση σωματικής βίας επίσης. 12 με 50% των γυναικών είναι θύματα σε βίας. Το οικονομικό κόστος της βίας κατά των γυναικών, και πάλι εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για 228 δις ετησίως, 45 δις σε απώλεια οικονομικής απόδοσης και τα υπόλοιπα ε, δίνει το κόστος ε, δηλαδή ουσιαστικών μέτρων είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος της βίας της ίδιας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει για, τη δημιουργία, για την πρόταση μάλλον μιας οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ήδη από το 2009 αλλά και το 2010 την ημέρα, ε, μάλλον καθιερώθηκε η ημέρα κατά της βίας ε, κατά των γυναικών εδώ. Επίσης υπήρξε μια νέα προσέγγιση για την καταπολέμηση της βίας μαζί με ποινικό δίκαιο. Το 2012 ε, εμείς ε, μέσα στην έκθεση της κυρίας Ιντεβέλτα ε, ζητήσαμε την παρουσία σε πολλές επιτροπής μιας ευρωπαϊκής, πανευρωπαϊκής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει και μέσα ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σήμερα υπάρχουν διάφορα μέτρα για να προωθούνται οι δράσεις στα κράτη-μέλη στον τομέα της πρόληψης της βίας, όμως δεν είναι καθολική η η στρατηγική. Ε, Τα επίπεδα προστασίας γυναικών και κοριτσιών κατά κάθε μορφής βίας διαφέρουν ε, στα κράτη-μέλη. Υπάρχει απουσία κοινής κατανόησης του ορισμού και των διατάξεων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στα διάφορα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζονται ελάχιστες προδιαγραφές, κοινή ορισμή, κοινή δράση για να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών και να εξασφαλίσουμε πως το πάνω από το ίμιση του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα χαίρει του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ένωση. Ένας κανονισμός είναι το καλύτερο μέσο ε, για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Δεν χρειάζονται εφαρμοστικά μέτρα και καθίσταται άμεσα ε, νόμος σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, θέμα είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις δράσεις των κρατών μελών ε, στον τομέα της ε, βίας κατά των γυναικών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες αλλά και κατάρτιση, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, συνειδητοποίηση του προβλήματος και ούτω καθεξής. Τώρα, στον τομέα της, το νομοθετικό, προτείνω καταρχήν η Κομισιόν μέχρι τα τέλη του 2014 να υποβάλει μια πρόταση για μέτρα για την προώθηση και στήριξη των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών. Δεύτερον, επιμένουμε για ένα συνεπές σύστημα για συλλογή στατιστικών όσον αφορά τη βία, την έμφυλη βία στα κράτη-μέλη. Ε, επίσης θα πρέπει να υιοθετηθεί με ομόφωνη απόφαση ε, συγκεκριμένοι ορισμοί θα ε, να προτείνουμε στην Κομισιόν να προτείνει ένα, ε, πρόγραμμα δράσης για την ε, βία κατά των γυναικών και να ξεκινήσει τη διαδικασία για την πρόσβαση της Ένωσης στα ίδια μέσα από τη στιγμή που θα έχει αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών. Επιπλέον, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν να, να προχωρήσει στα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη βία κατά των γυναικών, όπως, που θα είναι αντίστοιχο του Ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων. Επίσης, θέλουμε να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό έτος για την ε, κατάργηση της βίας ε, κατά των γυναικών με στόχο να αυξήσει την συνείδηση των πολιτών για το θέμα αυτό. Τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη η πρακτική της βίας δεν θα πρέπει να γίνεται πλέον ανεκτή και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει τον ηγετικό κανό, ε, μάλλον τον πρωτοπόρο ε, στην σχετική νομοθεσία και να ε, χρησιμεύσει ως παράδειγμα για όσους ε, νομικά, πολιτιστικά αλλά και πολιτικά προωθούν τη βία κατά των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος είναι λοιπόν στα μέλη μας, εάν θέλουν να σχολιάσουν τα όσα άκουσαν. Η κυρία Γκαρσία Πέρες είναι η πρώτη στον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί σε πολλές ε, περιπτώσεις για το θέμα αυτό νομίζω ότι περισσεύουν τα λόγια. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε με όλες τις σκέψεις της κυρίας Παρβάνοβα και θα ήθελα επιπλέον να την ευχαριστήσω για το περιεχόμενο της έκθεσης που προσαρμόζεται απόλυτα πρώτα απ' όλα στα όσα συζητάμε εδώ και πολλές συνεδριάσεις και στις επίσημες συναντήσεις μας και στις άτυπες επαφές και βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να εκφέρει άποψη για το θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα ουσιώδες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξαντλήσουμε τους χρόνους, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να το εγκρίνουμε πριν τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Τώρα, για αυτή την κοινωνική πληγή που είναι ε, η βία κατά των γυναικών, χτες εορτάσαμε την ε, ημέρα κατά της εμφυλής βίας. Ακούσαμε πάρα πολλές απόψεις που συμπίπτουν και που αποδεικνύουν πως αυτό το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών εξαρτώνται από το γεγονός και προέρχονται από το γεγονός ότι ζούμε σε μια άνηση, ριζικά άνηση κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εγκάρσια εφαρμογή αυτής της πολιτικής εξίσωσης προστασίας των θυμάτων σε όλους τους κλάδους. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι οι εκπαιδευτικές και προληπτικές πολιτικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Μία ακόμα γυναίκα αυτό το Σαββατοκύριακο δολοφονήθηκε από ε, τον πρώην, πρώην σύντροφό της. 45 έχουν ήδη δολοφονηθεί φέτος. Και αυτή η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 12 φορές. Είναι ο πρώην σύζυγός της και είχε καταγγείλει πως δεν σεβόταν την εντολή απομάκρυνσης που του είχε δοθεί. Οπότε 12 φορές την πλησίασε και την τελευταία φορά τη σκότωσε. Νομίζω πως τέτοιες περιπτώσεις που κρύβονται πίσω από τις συζητήσεις που κάνουμε για τους αριθμούς, αυτές οι ζωές που χάθηκαν, αυτές οι οικογένειες, τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, τα οποία έμειναν ορφανά, ε, είναι πολύ πιο ζωντανά από τους κρύους αριθμούς που εμείς συλλέγουμε. Θέλω λοιπόν να μην αναφερόμαστε μόνο στο κόστος της πολιτικής αυτής, γιατί ποτέ δεν θα επενδύσουμε αρκετά. για να μπορέσουμε να ξαπεράσουμε αυτή την πληγή. Γιατί και ένα μόνο θύμα να δολοφονηθεί από πρώην σύντροφο, επειδή ακριβώς είναι γυναίκα, θα έχει φανεί πως κανένας προϋπολογισμός και κανένα, καμία πρικοδότηση από τις κρατικές υπηρεσίες δεν είναι επαρκής είτε είναι εθνική η χρηματοδότησή τους είτε κοινοτική. Ελπίζω λοιπόν οι συζητήσεις αυτές οι οποίες γίνονται βασιζόμενες σε εκθέσεις δεν θα μείνουν στα λόγια αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια εδώ όλα τα ευρωπαϊκά όργανα για να προχωρήσουμε σε αυτή την μάχη κατά αυτής της κοινωνικής πληγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματέρα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ παίρνω το λόγο στο όνομα της Κιόδους για το ΕΛΚ που είναι η κυρία Τερέζα Χιμένας και που σήμερα δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ ε, λόγω θεσμικών υποχρεώσεων. Θα διαβάσω το σημείωμα που μου έστειλε προσωπικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παρβάνοβα που τονίζει τη σημασία καταπολέμησης τη βία κατά των γυναικών. Θεωρώ πως είναι πλήρης η εκθέση τη που καλύπτει όλες τις πτυχές τη βία κατά των γυναικών. Έχω την πρόθεση να υποβάλω κάποιες τροπολογίες που στόχο έχουν να τονίσουν τη σημασία των θυμάτων τη βία κατά των γυναικών που συμπεριλαμβάνουν ανήλικε ε, ε, τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων ε, εμπόριο ε, κομματιών του ανθρώπινου σώματος και ούτω καθεξής. Το μόνο πρόβλημα που συνάντησα σε αυτή την έκθεση αφορά το άρθρο 3 το οποίο ζητά τον να γίνει εντοπισμό κατά το, της κατά των γυναικών ε, και να θεωρηθεί ως έγκλημα στο πλαίσιο της παραγράφου 83 ε, τμήμα F. Νομίζω πως αυτό είναι σημαντικό ε, σημείο γιατί όντως καταπολεμάται έτσι η βία. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Παρβανόβα πώς θεωρεί, ποια θεωρεί ότι θα είναι τα προβλήματα που θα συναντήσουμε σε αυτό το, πεδίο, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τροποποιήσουν τις εθνικές νομοθεσίες σε περίπτωση που αυτή εδώ η ε, πρόταση γκριθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέρτμαν μετά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θεωρώ εξαιρετική την έκθεση, έτσι όπως είναι. Και θεωρώ επίσης εξαιρετικά λυπηρό ότι σήμερα συζητούμε ένα τέτοιο θέμα. Η γυναίκα είναι και αυτή άνθρωπος. Ο άνδρας είναι άνθρωπος. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν ένας άνδρας συμπεριφέρεται έτσι σε έναν συνάνθρωπο. Δυστυχώς πάντα και, και στη δική μου χώρα ισχύει αυτό, πάντα πρέπει να συμβεί κάτι μέχρι να πάρουμε στα σοβαρά μια κατάσταση. Και έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους και μαθαίνω ότι έγινε κάτι και μετά υπήρξε αντίδραση. Και γίνονται πράγματα, δεν τα παίρνουμε στα σοβαρά και μετά όταν η κατάσταση φτάνει στο μη περαιτέρω καλούμαστε να κάνουμε κάτι. Γιατί τόσο αργά. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και το σχέδιο δράσης, πιστεύω πως είναι εξαιρετικό, πως είναι τέλειο, το στηρίζω απόλυτα, όμως ε, ζητώ τα κράτη-μέλη να φροντίσουν έτσι ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη και να μην μείνουν στη θεωρία αυτά που αναφέρεται στην έκθεση. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Νομίζω πως η έκθεση είναι καλή γιατί κανείς δεν, μπορεί, δεν περισσεύουν καθόλου λόγια για αυτή του είδους βία. Εκεί θα πρέπει η ανοχή να είναι μηδενική. Όμως, γιατί πάντα στη ζωή μου εγώ έχω ένα όμως. Ανησυχώ για το γεγονός ότι θέλουμε να νομοθετήσουμε και άλλο. Δεν νομίζω ότι περισσότερη νομοθεσία είναι πάντα ο τρόπος για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένη δράση και θα πρέπει στην αιχμή αυτής της δράσης να είναι τα κράτη-μέλη, να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές, να δούμε τι έχει λειτουργήσει στις διάφορες χώρες. Να σας εξηγήσω λοιπόν τι γίνεται ε, με μια περίπτωση με την οποία ασχολούμαι αυτή την εποχή. Ήταν παιδιά που πήγανε διακοπές στην Ελλάδα και βιάστηκαν και ο τρόπος που τις μεταχειρίστηκαν οι αρχές ήταν αειδιαστικός. Εγώ το παρακολουθώ. Η νομοθεσία υπάρχει. Οι αρχές δεν ήξεραν πώς να την εφαρμόσουν και δεν την εφήρμοσαν σωστά. Αυτή τη στιγμή μιλώ με ομάδες στήριξης θυμάτων βιασμού και στις δύο χώρες για να δούμε τι θα κάνουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι πιο συγκεκριμένο, όχι μόνο νομοθεσία και πάλι νομοθεσία. Θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι να συνεργαστούν και να συντονίσουμε τις δράσεις μας και θα το κάνουν. Τώρα για τα στατιστικά στοιχεία, ωραία να συλλέξουμε και άλλα. Λοιπόν, αξίζουν, γιατί πολλές φορές η βία δεν καταγράφεται όσο θα έπρεπε. Τώρα, για τον μηχανισμό που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, και για το θέμα των ακροτηριασμών με τον οποίο εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ, θέλω να δω πώς μπορούμε να έχουμε την αιρεσιμότητα ε, στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρουμε σε χώρες οι οποίες προχωρούν σε ε, τέτοιου είδους ακροτηριασμό και δεν είμαι καν ήδη Μήπως θα έπρεπε να σέβονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, οι κυβερνήσεις πριν λάβουν αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν μιλώ για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και για τα κριτήρια της Κοπενχάγης ρωτώ το εξής. Εκεί δεν λέμε πως τα κράτη-μέλη στο κριτήριο της ισότητας έχουν πολιτική για να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο νομοθεσία. Ε, thanks for that. Ε, we have... Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Τρεις ομιλητές παραμένουν. Μετά θα κλείσω τη συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Κλεβέτη. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που αργοπόρησα, ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να ψηφίσω σε άλλη επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο μου σχόλιο έχει να κάνει με την ε, ερώτησή μας ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ερώτηση την οποία συνυπογράψαμε πολλοί ευρωβουλευτές για την ανάγκη και το πότε θα κυρωθεί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη ερώτηση αυτή. Και δεύτερη, δεύτερο σχόλιο μάλλον, θα ήθελα να τονίσω το ότι η οδηγία ε, για την περιοριστική εντολή ήδη έχει καθυστερήσει τρία χρόνια. Στα τρία αυτά χρόνια τα κράτη-μέλη έπρεπε να κυρώσουν και να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία την οδηγία για την περιοριστική εντολή. Εμείς ως Επιτροπή αρμόδια για αυτό το θέμα, για το θέμα της έμφυλης ε, βίας, θα πρέπει να ελέγχουμε την πρόοδο της μεταφοράς της οδηγίας από τα κράτη-μέλη στην εθνική νομοθεσία. Πρέπει να το θεωρήσουμε έναν στόχο μας για τις μελλοντικές μας δραστηριότητες. Τρίτον, όσον αφορά την ίδια την έκθεση, φυσικά και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση και συγχαίρω την ε, Αντωνία γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμως, να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή μας έχει και άλλη μια έκθεση. Ε, την έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ για την πορνεία. Και στην έκθεση αυτή γίνεται λόγος για την ε, πορνεία ως μορφή έμφυλης βίας. Ίσως λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή. Σίγουρα αυτή είναι μια νέα ιδέα της έκθεσης της κυρίας Παρβανόβα. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε την προηγούμενη έκθεση, αν συμφωνεί βέβαια και η Αντώνια, και να την συνδυάσουμε και να, μπορού, και να θεωρήσουμε ενδεχομένως την πορνεία ως μια μορφή ε, βίας κατά των γυναικών και σε αυτήν την έκθεση έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ πιο δυνατή έκθεση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα θέμα συνοχής. Εγώ προσωπικά θα συνεισφέρω με τροπολογία στην έκθεση αυτή και ελπίζω να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα για τις γυναίκες, για τα θύματα αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Κράτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητούμε και πιστεύω ότι όλοι συμμετέχουμε με μεγάλη προσοχή και προσήλωση. Ε, θέλω να αναφερθώ στην αναφορά της κυρίας Γιανακουδάκη για τις βιασμούς των παιδιών στην Ελλάδα από ό,τι αντελήφθηκα. Ε, φαντάζομαι ότι κάπου θα βασίζεται η κυρία Γιανακουδάκη. Ήθελα μόνο να τη ζητήσω κάποια στοιχεία διότι ε, ξέρετε η ελληνική κοινωνία είναι πολύ αλληλέγγυα από τα παιδιά και το παιδί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, κουλτούρα και στην κοινωνία μας και οι παρατυπίες που η σοβαρή παρατυπία που εξέφρασε η κυρία Γιανακούδακη μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα να τη ζητήσω στοιχεία από αυτού. Ευχαριστώ. Ε, ε, κυρία Γιανακουδάκη, έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Ευχαριστησή μου. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά. εξασκήσω τα αγγλικά μου. Αναφέρομαι λοιπόν σε δύο κορίτσια τα οποία πήγαν να ζήσουν στην Ελλάδα για ένα χρόνο πριν τις σπουδέ τους και βιάστηκαν ομαδικά αφού πρώτα τους ε, δόθηκαν ναρκωτικά. Το πρόβλημα ήταν η μεταχείριση από την αστυνομία και ο τρόπος ε, με τον οποίο έγινε αυτό. Πήγαν στην αστυνομία και τους ε, είπαν να επιστρέψουν την επόμενη μέρα για να κάνουν κατάθεση, να μην ε, πληθούν, να συλλέξουν τα αποδεικτικά στοιχεία από το διαμέρισμά τους σε πλαστικές ε, σακούλες, δηλαδή να μολύνουν με τα δικά τους αποτυπώματα τα αποδεικτικά στοιχεία και εγώ προσωπικά πήγα στην Ελλάδα πριν από περίπου ένα μήνα. Ε, τα κορίτσια αυτά έδωσαν συνέντευξη στην καναδική τηλεόραση γιατί είναι ελληνοκαναδέζες και με τα χαρά μου να μοιραστώ τις πληροφορίες και ίσως κάνουμε κάτι μαζί για το θέμα αυτό. Τέλος, ο υποφαινόμενος. Είμαι σκιώδης εισηγητής και με αυτή την ιδιότητα θα μιλήσω. Θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η έκθεσή σας, κυρία Παρβάνοβα, είναι εξαιρετική. Και χαίρομαι πολύ που τώρα τονίζουμε το σημείο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μία οδηγία για την έμφυλη και για πάρα πολλούς λόγους χρειάζεται και είναι υπεύθυνη και είναι αναγκαία μια τέτοια νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες κάθε μέρα υπόκεινται σε έμφυλη βία. Η βία όμως αυτή είναι και μια άμεση αντανάκλαση της πατριαρχικής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Και από εκεί παίρνει και την έκταση που έχει πάρει. Χρειάζεται λοιπόν να ορίσουμε την έμφυλη βία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφανθεί για το τι θεωρεί έμφυλη βία. Το κάναμε αυτό στην έκθεση Σβένσον το 2011, όπου συμπεριλαμβάνουμε όλα τα συστατικά στοιχεία, όλες τις συνιστώσεις της έμφυλης βίας συμπεριλαμβανόμενης και της πορνείας. Πέραν αυτού, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία της έκθεσης, τα οποία θεωρώ πως είναι εξαιρετικά, κυρία Παρβάνοβα, και σε κάποια άλλα πράγματα, τα οποία ίσως να ξαναδούμε και να συζητήσουμε. Πιστεύω πως το σημείο 4 είναι εξαιρετικό, όπου ζητείται από τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι μια εξαιρετική σύμβαση που δημιουργεί ε, ισχυρά και γερά πρότυπα και πιστεύω πως όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να κυρώσουν την σύμβαση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι τονίζεται η θέσπιση ενός έτους αφιερωμένο στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το πόσο σημαντική είναι αυτή η μήνυ οδηγία. Τα κράτη-μέλη χρησιμοποιώντας την αρχή της επικουρικότητας θα μπορούν να βρουν τους ε, καλύτερους δυνατούς τρόπους εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Τώρα, ε, με για το αντίθετο, αλλά νομίζω πως υπάρχει ήδη ένας ορισμός για το τι καθιστά εμφυλιβία. Δεν βλέπω την ανάγκη να ορίσουμε και εδώ την, τον ακροτηριασμό των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων ως συστατικό στοιχείο της έμφυλης βίας. Επίσης πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είναι αδρανής, αλλά απλά έχει επιλέξει ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτές τις μορφές ως μέρη ενός συνόλου άλλων εκφάνσεων εμφυλής βίας. Έπειτα, δεν είμαι, σίγουρη, δεν είμαι σίγουρος εάν ξεπερνά τα, τα όρια της έκθεσης αυτής. Αλλά υπάρχουν οργανώσεις γυναικών οι οποίες εμάχονται εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να έχουν την επαρκή χρηματοδότηση και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης όπου τα κράτη-μέλη δεν έχουν πόρους, όπου οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν πόρους. Ταυτόχρονα αυξάνονται τα κρούσματα βίας, ενώ οι οργανώσεις αυτές δεν διαθέτουν τους πόρους για να ε, δράσουν, για να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενο αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εσείς κυρία Παρβάνοβα το τονίζετε. Τονίζετε τη σημασία των οργανώσεων ε, αυτών. Και ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την ε, ανάγκη ύπαρξης ενός ειδικού εισηγητή. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα σημεία ήθελα να θίξω. Κατά τα άλλα είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την έκθεση αυτή και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε και να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή πριν το τέλος της εθιτείας μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτό. Τώρα, θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μπανκέ ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στις ερωτήσεις της ε, κυρίας Εκλεβέτη και της ε, κυρίας Γιανακουδάκη που έχουν να κάνουν με την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα θα ήθελα να ρωτήσω αν η, κυρία, η εκπρόσωπος της Επιτροπής θα ήθελε να λάβει το λόγο. Um, yes, thank you very... Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για το σχέδιο έκθεσης. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερο το κείμενο αυτό και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Βαρβάνοβα που το κατέθεσε γιατί μιλάει με πολύ ε, ένταση για την δέσμευση που έχουμε αναλάβει όλοι να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Είναι μια δέσμευση λοιπόν και της εισηγήτριας και της δικής σας επιτροπής για το θέμα της βίας κατά των γυναικών αντιμετωπίζοντας τις ε, πραγματικές αιτίες αυτού του φαινομένου. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μοιραστούμε αυτή τη δέσμευση για να το πετύχουμε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες ήταν η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και εγκρίθηκε μια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης για, τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών και είναι η πρώτη φορά που μίλησε με τόσο απερίφραστο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσίασε συγκεκριμένες δράσεις που έχουν να κάνουν και με την εταιρική σχέση με τις οργανώσεις που επιτόπου συνεργάζονται και με τα θύματα αυτό το ακροτηριασμού και με τα ενδυνάμει θύματα. Και μαζί τους φτιάξαμε και το σχέδιο δράσης και την ανακοίνωση έτσι ώστε να γίνει μια δράση πρόληψης προστασίας των θυμάτων και των ενδυνάμει θυμάτων όπως επίσης και η δίωξη των αυτούργων. Για ένα από τα θέματα τα οποία ανέφερε η συγγήτρια, που είναι το σχέδιο δράσης για τον ε, γενετικό ακροτηριασμό των γυναικών, πρέπει να σας πω πως περιμένουμε με μεγάλη προσδοκία τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Επίσης, να σας πω πως πολλά από τα σχόλια που ακούστηκαν και που βρίσκονται στο σχέδιο έκθεσης, τα στηρίζουμε απόλυτα. Τα έθιξαν δε και άλλα ε, μέλη της Επιτροπής σας. Πρώτα απ' όλα, η ανάγκη να έχουμε ε, στοιχεία στα οποία να μπορούμε να βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βία κατά των γυναικών. Δεν έχουμε ακόμα αρκετά αξιόπιστα στοιχεία. Θα πρέπει να μετρήσουμε και τη διάσταση του φαινομένου και τον αντίκτυπο που έχουν όλα τα είδη βίας κατά των γυναικών. Mm. Αναμένουμε λοιπόν με χαρά την πρώτη ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή έρευνα για την βία που θα παρουσιάσει η οργάνωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα του χρόνου. Επίσης θέλουμε να δούμε τι θα πει και το Ινστιτούτο στο Βίλνιος για την ισότητα μια που έχει και αυτό ρόλο να παίξει στη συλλογή των στοιχείων και στην βελτίωση των ποιοτικών στοιχείων που έχουμε Θα ζητήσουμε από το Ίδρυμα αυτό να ανεβάσει ρυθμούς για τη συλλογή δεδομένων και με χαρά βλέπουμε πως την έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνουμε τα ίδια στοιχεία που θα επιτρέψουν ε, να λάβει δράση το συντομότερο. On the importance of awareness. Επίσης συμφωνούμε για το πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού ε, για την ε, βία κατά των γυναικών και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι ολοκληρώσαμε τις διαβουλεύσεις ε, για να ενισχύσουμε την χρηματοδότηση σε εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού κατά της έμφυλης βίας για τα επόμενα δύο χρόνια και προβλέπουμε επίσης ε, χρηματοδότηση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια κονδύλια τα οποία θα δοθούν σε αυτές τις 14 εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Πέραν από την ε, δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε, θα συνεχίσουμε μάλλον να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Δάφνη και να συνεργαζόμαστε με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται κατά της ευβίας και όλων των εκφάνσεων της. Τώρα, όσον αφορά την νομοθεσία... Η Κομισιόν ε, πρότεινε ένα πακέτο για τα θύματα, το οποίο έχει εγκρίθει, που βασίζεται κυρίως στις προσπάθειες ε, που γίνονται για τα θύματα, που, για τις γυναίκες που έφτουν θύματα έμφυλης βίας και στοχεύει πιο ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία στήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για το πώς θα γίνει η μεταφορά αυτής της οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία και ποια θα είναι η σωστή και συνολική εφαρμογή αυτής. Όταν μιλάμε για νέα νομοθεσία για τη βία κατά των γυναικών, τα θέματα τα οποία προκρίνονται από το σχέδιο έκθεσης θα πρέπει να αναλυθούν με λεπτομέρειες από τους ε, νομικούς μας, γιατί υπάρχει και το θέμα της νομικής βάσης και το κατά πόσο χρήζει η μορφή να είναι κανονισμός. Όταν όμως διάβασα τα όσα είπε η συγγήτρια για το τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει η οδηγία και πάλι αναφέρθηκε πως πρέπει να ανταλλάξουμε εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές, να οργανώσουμε επιμόρφωση, συγκέντρωση στοιχείων, ευαισθητοποίηση, στόχοι λοιπόν τους οποίους προσυπογράφουμε. Και βέβαια είναι θέματα τα οποία όχι μόνο συζητάμε, αλλά και για τα οποία παραδίδουμε από τα αποτελέσματα. Θα κλείσω εδώ. Είναι εξαιρετικά επικοδομητική έκθεση. Βεβαίως οι λεπτομέρειες θα πρέπει, ή τουλάχιστον η νομική τους διάσταση, να εξεταστούν περαιτέρω. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια για το σχέδιο αυτό που έχει καταθέσει. Ευχαριστώ. Μπορείτε λοιπόν να απαντήσετε και στα όσα είπε η συνάδελφος για το που βρισκόμαστε στη διαδικασία για την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία καλύπτει σε μεγάλο βαθμό εθνικές αρμοδιότητες, δηλαδή τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Και η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ που είναι η Επίτροπος η Αρμόδια δεν ξεχνά σε καμία περίπτωση να υπενθυμίσει στα κράτη-μέλη να κυρώσουν. Μόνο η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν επικυρώσει μέχρι σήμερα. Εμείς πιέζουμε τα κράτη-μέλη να την επικυρώσουν, η οποία είναι και σημαντική και σφαιρική. Αυτή τη στιγμή σε εσωτερικό επίπεδο να λύουμε ποιες είναι οι νομικές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει ως μέλος. Είναι και αυτό μια δυνατότητα που άνοιξε η Σύμβαση, όπως επίσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ακόμα πάντως δεν έχουμε αποκτήσει αρκετή εμπειρία. Πρόκειται δηλαδή για μια πρόσφατη ε, δυνατότητα να προσχωρεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος ε, σε ε, διεθνείς συμβάσεις και θέλουμε να δούμε οι επιπτώσεις ποιες θα ήταν σε νομικό επίπεδο. για να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας και τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης του επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Συγχωρέστε με. Δεν θέλω να είμαι αγενής. Αλλά πείτε μας πόσο θα χρειαστείτε για να το αναλύσετε. Γιατί έχετε καιρό που αναλύετε. Κατανοώ πως αντιμετωπίζετε προβλήματα και υπάρχουν και νομικά κολλήματα, αλλά έχετε κάποια πρόβλεψη να κάνετε για το χρονικό ορίζοντα. Τι να σας πω, τι προβλέπω. Τους επόμενους μήνες για κάποια αποτελέσματα. Κατανοήστε όμως και εσύ πως η σύμβαση αυτή καλύπτει εθνικές αρμοδιότητες δεν υπάρχει ούτε ένας κανόνας στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης για την οποία την αρμοδιότητα φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αποκλειστικό τρόπο. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη πρέπει να επικυρώσουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Συμφωνώ. Συμφωνώ και αυτό εξετάζουμε. Πώς θα μπορούσε να έχει μια προστιθέμενη αξία η προσχώρηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αναλύουμε. Και ελπίζουμε στους επόμενους μήνες άντε αρχή της επόμενης χρονιάς να έχουμε κάποια από τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κυρία Κλεβέτη, πολύ σύντομα. Ίσως είναι νομικό το ζήτημα, αλλά παράλληλα στο κείμενο της σύμβασης, της ε, σύμβασης Κωνσταντινούπολης γράφει. Γιατί μιλάμε για έγγραφο το οποίο ήδη υπάρχει, πως είναι ανοιχτό σε κύρωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι λοιπόν πως η, νομική η νομική υπηρεσία εκεί έχει αναλύσει την κατάσταση και θα ήταν εξαιρετικό το μήνυμα προς τα κράτη-μέλη για να τα οθήσει προς την κύρωση αυτή, να δούμε πως τουλάχιστον έχουμε γνωμοδότηση θετική της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να πει ναι, θα προχωρήσουμε κι εσείς θα δούμε το πρόβλημα και ενδεχομένως θα προχωρήσουμε και εμείς σε κύρωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολύ λίγα κράτη-μέλη έχουν κάνει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Πρέπει να πιεστούν. Ε, ενδεχομένως μέσω τέτοιας γνωμοδότησης. Δεν λέω πως αύριο θα έχει τελειώσει το θέμα της κύρωσης, αλλά τουλάχιστον αυτή η προσέγγιση, το μήνυμα. Θα ήταν χρήσιμο νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η συγγήτρια κυρία Παρβανόβα για τα τελευταία σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ όλους όσους ε, διατύπωσαν την άποψή τους και έκαναν προτάσεις. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του με τη μορφή τροπολογιών, αν και δεν έχουμε μεγάλη χρονική προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. Συζητούμε πολύ καιρό την έκθεση αυτή. Ε, οι προθέσεις τη επιτροπή είναι ξεκάθαρες και οι συνάδελφοι έχουν ήδη ετοιμάσει τις τροπολογίες τους. Τώρα, να απαντήσω στην ε, κυρία Ματέρα και στην ε, απόψη της για το άρθρο 83 παράγραφος 1 ότι η έμφυλη βία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ε, ρήτρα παρέκτασης. Να τη υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με την ρήτρα αυτή ε, απαιτείται ομόφωνη απόφαση για το αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και μια άλλη μορφή εγκλήματος. Όμως θεωρώ πως ε, υπάρχει κάποιος συνδυασμός ε, και υπάρχουν διαφορές στις ε, μορφές αυτές. Κάποια εγκλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά, κάποιες μορφές έχουν κοινωνικό, οικονομικό χαρακτήρα. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν αυτή την πρόταση, διότι έχουμε πολύ ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά το πόσο αριθμό μεγάλος αριθμός γυναικών έχει επηρεαστεί. Νομικές συνέπειες ε, έχει αυτό. Υπάρχει και, μια, υπάρχει και αντίστοιχη μελέτη, αξιολόγηση για την ευρωπαϊκή Προσθέμενη αξία. Έπειτα. Η έκθεσή μας ε, υποστηρίζει την ε, συμπερίληψη της έμφυλης βίας και του προβλήματος αυτού στο πεδίο εφαρμογή Φυσικά εδώ συμπεριλαμβάνεται η τομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, η διακίνηση ε, ανθρώπων. όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη ρήτρα παρέκτασης. Όμως έχουμε επίσης εκτός από αυτά και την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, τα οποία εξετάσαμε εκτενώς, επίσης την ε, το ξέπλυμα χρήματος, την διαφθορά, το κυβερνοέγκλημα, τα οποία πιστεύω πως δεν έχουν καλυφθεί αρκετά από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεδομένου ότι η νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες και η διαφθορά είναι κάτι που είναι πράγματα που αξίζουν περισσότερη προσοχή από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεν καλύπτονται παρκώ από την νομοθεσία, δεν βλέπω λόγο να μην συμπεριληφθεί σε αυτά και η έμφυλη βία, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη ε, ε, ιστορία και πάει πολύ πιο πίσω από ότι το ξέπλυμα χρήματος. Και έχει και σοβαρό αντίκτυπο οικονομικό και κοινωνικό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να συμπεριληφθεί αυτή από τα κράτη-μέλη. Τώρα όσον αφορά την πορνεία. Καταρχάς, ακριβώς επειδή προτείνουμε νομοθεσία και ορισμούς, παραπέμπουμε στον ορισμό την στήριξη των θυμάτων, την αντίστοιχη οδηγία και παραπέμπουμε και στους διεθνείς ορισμούς που χρησιμοποιεί ο ΙΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Καταρχάς ε, συμφωνείτε ότι η πορνεία θεωρείται έγκλημα και όχι μόνο έγκλημα αλλά ε, βία κατά των γυναικών και μορφή διάκρισης και αυτό πρέπει να φανεί και στι τροπολογίε τώρα όσον αφορά τον ακροτηριασμό των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων. Χρησιμοποιούμε τον ακροτηριασμό διότι ήδη υπάρχει μια μελέτη, ήδη υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράση για αυτό. Και φυσικά και υπάρχουν και άλλες μορφές βίας κατά των γυναικών, όμως η αναφορά στον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων θα είναι μια θετική εξέλιξη όσον αφορά την ενίσχυση της διασωνοριακής διάσταση και της εξωτερικής διάστασης της έμφυλης βίας. Τώρα, όσον αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε. Και χαίρομαι πολύ που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επένους για τον ε, ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τώρα, οι πόροι πιστεύω πως ε, πρέπει να διατίθενται με συνεκτικό τρόπο και να έχουν συνέχεια και να υπενθυμίσω και ότι σε αυτή την επιτροπή το παλεύουμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Πρέπει να στηρίζεται οικονομικά. Γι' αυτό προτείνω να μην αφαιθεί στην πολιτική θέληση. Πρέπει να στηριχθούν οικονομικά οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που προσπαθούν να καταπολεμήσουν και να ευαισθητοποιήσουν για τη βία κατά των γυναικών. Ας μην το βάλουμε σε ψηφοφορία λοιπόν. Τέλος, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αληθεύει ότι η Πορτογαλία στηρίζει τη σύμβαση, έχει προσχωρήσει, όμως δεν ε, συμφωνώ με μία αρχή της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει τις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και εάν υπάρχουν τουλάχιστον 8 κράτη-μέλη που συμφωνούν, πρέπει να θεωρηθεί μια νέα πρόταση και να έχει μια βαρύνουσα σημασία. Και μετά από διαβουλεύσεις μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, να πω ότι λάβαμε ήδη ορισμένε θετικές απαντήσεις όσον αφορά την διαδικασία κύρωσης από τη Φιλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία, πέραν από την Ιταλία και την Πορτογαλία. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη που θα έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις και, θα συμβάλλει σημαντικά ώστε να γίνει νομοθετική πρόταση. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ξανά όλους όσους έχουν συνεισφέρει και να σας υπενθυμίσω ότι προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι πολύ σύντομη, Δυστυχώ, λυπάμαι γι' αυτό, είναι αύριο στι 5 το απόγευμα. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, δεχτείτε τη συγγνώμη μου για αυτήν την σύντομη προθεσμία. Ο λόγος ε, που λίγη αύριο είναι ότι θέλουμε να την ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Μάρτιο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Δεν θέλω ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να, να αναβληθεί για τον Απρίλιο και να υπάρξει ενδεχόμενο να περάσει στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παρβανόβα. Ως πρόεδρος ε, είμαι υποχρεωμένος να σας επαναλάβω την προθεσμία για τις τροπολογίες. Η Αντώνια ήδη τις ανέφερε, αλλά θα τις πω και εγώ άλλη μια φορά. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών αύριο 27 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στις 6 Δεκεμβρίου, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή τον Ιανουάριο και η έκθεση θα πάει στην Ολομέλεια μάλλον το Μάρτιο. Μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και να πω ότι υπάρχουν αντίγραφα της μελέτης που σας παρουσιάστηκε νωρίτερα ε, έξω από την αίθουσα. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε ένα αντίγραφο φεύγοντας. Προχωράμε όμως στο σημείο 13 της ε, μετανάστριας χωρίς ε, ε, επίσημα έγγραφα. Να σας πω ότι επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, θα εκτιμήσω πολύ την συντομή παρουσίασή σας. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο. Στη... Κανονικά θα έπρεπε να δώσω το λόγο στην κυρία Νικολάη, η οποία πουσιάζει στην κυρία... Μετά η αντικαταστάτριά της ήταν η κυρία Ολυβία, η οποία επίσης απουσιάζει και θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα, η οποία θα μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Και να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μιλήσετε μπορείτε να πάτε έξω. Εδώ πρέπει να κάνετε ησυχία. Κυρία Παρβανόβα. Επειδή εγώ έχω έρθει για να αντικαταστήσω την κυρία Νικολάη που είναι σε αποστολή και την κυρία Σέρ που είναι σε άλλη βιτροπή και ψηφίζει, θα σας διαβάσω απλώς αυτά τα οποία θέλει να συμπεριλάβουμε η κυρία Νικολάη και το οποίο απευθύνει σε εσά. Αγαπητοί συνάδελφοι, λυπάμαι ιδιαίτερα που δεν είμαι σε θέση να παρευρεθώ σήμερα να υποβάλω τη δήλωση αυτή. Είμαι σε αποστολή στην Αιθιοπία. Σας ευχαριστώ όλους που υποβάλατε τόσο ε, σχετικές ε, τροπολογίες, τις διάβασα προσεκτικά και πιστεύω πως μπορούν να στηριχθούν σε μεγάλο βαθμό. Θα υποβάλω συμβιβαστικές τροπολογίες, τις οποίες το γραφείο μου θα σας στείλει σύντομα. Επίσης, ενδεχομένως θα γίνει μια σύντομη συνεδρία των ε, σκιωδών πριν συναντηθεί και πάλι η Επιτροπή μας 16 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Ματέρα είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ παίρνω το λόγο ως σκιώδης για αυτή την έκθεση για το ΕΛΚΑ. Είναι βεβαίως μια έκθεση που αγγίζει ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το θέμα των ε, μεταναστριών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για γυναίκες που δεν μπορούν να έχουν κοινωνική αρρωγή ούτε υγειονομική περίθαλψη. Είναι γυναίκες που ωστόσο πολύ συχνά Ε, αποτρέπονται από το να κάνουν καταγγελίες αν είναι θύματα καταχρήσεων ή βίας. Γι' αυτό και ε, συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τη θέση της συναδέλφου Νικολάη, κυρίως όσον αφορά την εκμετάλλευση των γυναικών στον κόσμο της εργασίας ή και στον κόσμο των ε, ε στις στα σπίτια όπου αυτές διαμένουν, δηλαδή είναι πιο ευάλωτες. Η έκθεση εισάγει συγκεκριμένες ε, καινοτομίε Έχω συμμετέχει με, και έχω διαβάσει 69 τροπολογίε που υπευλήθησαν, αλλά υπογραμμίζω κάποιε που κατά τη γνώμη μου ήταν κάπως εκτό θέματο. Όπω α πούμε οι 37 ή κάποιες άλλες που ήταν πολύ γενικόλογες, 18-24, αλλά με πάση περιπτώσει η κάποιε άλλε που ηταν πολυ γενικολογες 18 24 αλλα με παση περιπτωσει η συναδελφο δεν είναι παρούσα. Ίσως λοιπόν θα έρθω σε επαφή μαζί τη και θα τη δώσω τι γραπτέ μου σημειώσει για να κάνουμε μια σύγκριση γιατί πιστεύω η κυρία Παρβάνοβα δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό αφού απλά διαβάζει εξ ονόματος των συναδέλφων κάποια έγγραφα. Άρα λοιπόν είναι άσκοπο να συνεχίσω να λέω τις λεπτομέρειες γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορώ να το συζητήσω με την εισηγήτρια σήμερα. Έχω πιο συγκεκριμένε παρατηρήσει να κάνω, οπότε να πω εν γέννη πω εγκρίνω αυτή την έκθεση, τη στηρίζω και μαζί με το ΕΛΚΑ σίγουρα θα συνεργαστούμε εξαιρετικά για ένα θέμα που είναι πολύ επίκαιρο και επίγον, γιατί υπό το φως των όσων συμβαίνουν στην Ιταλία, στη Λαμπεντούζα, με όλες αυτές τις αποβάσεις ε, μεταναστών, αυτές, αυτά τα ταξίδια, τις ελπίδες, αυτές οι γυναίκες που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους, ε, μας δίνουν ακόμα ένα επιχείρημα πως η Ευρώπη θα πρέπει να τη λάβει υπόψη κατά προτεραιότητα, γιατί είναι σαφές πως η ε, Ευρώπη είναι και η Λαμπεντούζα. Είναι η πιο νότια άκρη της Ιταλίας. Ε, πρόκειται για γυναίκες μετανάστες που θα πρέπει πραγματικά λοιπόν να αναλυφθούν υπόψη. Η συνάδελφος με δει λοιπόν ότι θα είμαι πολύ δραστήρια για αυτό το θέμα που εγώ προσωπικά ως εκπρόσωπος της Νότιας Ευρώπης είμαι πολύ ευαίσθητη σε όλα αυτά και θα είμαι ακόμη πιο δραστήρια. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια σύντομα γιατί είμαι και εγώ σκιώδης. Εδώ η πρόταση είναι καλή και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλω να καταθέσω και εγώ έχω μάλλον καταθέσει και εγώ κάποιες τροπολογίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, ε, ευαίσθητη κατάσταση στην οποία βρίσκονται την ευάλωτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μετανάστες όταν φτάνουν εδώ. Εκτίθενται σε εκεί βία, σε στην πορνεία, αλλά και τα κορίτσια και τα παιδιά δηλαδή ε, κινδυνεύουν εδώ. Καταρχήν είναι λοιπόν καλή η έκθεση, έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες και ελπίζω πως η συγγήτρια θα λάβει υπόψη τις τροπολογίες μου. Πιστεύω πως είναι καλές ή τουλάχιστον τις συμπεριλάβει σε συμβαστικές ε, μαζί με άλλες δηλαδή, σε συνδυασμό με άλλες. Να ρωτήσω λοιπόν αν κάποιος από την Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Yes, please, you have the floor. Yes, thank you, Chair. Very briefly. Ναι, πρόεδρε, πολύ σύντομα γιατί ξέρω πως δεν έχουμε χρόνο και όντως η συγκίτρια λείπει, οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Να κάνω δύο παρατηρήσεις ενημερωτικά όσον αφορά το πλαίσιο των κυρώσεων της κατάθεσης ανωνύμων καταγγελιών για τις μετανάστρες ε, ε, χωρίς έγγραφα που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το άρθρο 13 της οδηγίας δεν απογορεύει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν ανώνυμα ε, το τι τους έχει συμβεί. Αυτό που λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την ε, οδηγία διευκόλυνσης και αυτό αναφέρεται εδώ. Ίσως να είναι χρήσιμο ε, να διαπιστώσουμε πως η ε, Κομισιόν έχει κάνει μελέτη, είναι υπό εξέλιξη για ανημέρωση της μεταγραφής ε, του πακέτου διευκόλυνσης, όχι μόνο δηλαδή την Οδηγία 2002-90, αλλά και τη συμπληρωματική απόφαση πλαίσιο για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων της παράνομης μετανάστευσης δηλαδή. Ε, τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σε 6 με 8 μήνες, ώστε στόχος είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη μέσα στο 2014. Αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Έχουμε... Δεν έχουμε άλλον στον κατάλογο μιλητών. Μπορώ να σας πω το χρονοδιάγραμμα. Θα το ψηφίσουμε στις 16 Δεκεμβρίου και θα περάσει από την Ολομέλεια μάλλον το Φεβρουάριο. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση του σημείου 13 και περνάμε στο σημείο 14. Η διαχείριση της επιστροφής, συνεργασία με τρίτες χώρες, αποτελεσματική εφαρμογή συμφωνιών και πρακτική εφαρμογή της οδηγίας περί της επιστροφής. να δώσω το λόγο στην κυρία Ματέρα, από ό,τι φαίνεται, <laughs> όχι στην εισηγήτρια. Ναι, Πρόεδρε, εγώ λίγο αφαιρέθηκα. Νομίζω πως μιλάτε για την Ρόζα Εσταράς Φεραγκούτ. Ναι, α, με συγχωρείτε γιατί αφαιρέθηκα. Μάλιστα, παρούσα, παρούσα. Εδώ σήμερα είμαι η εισηγήτρια <laughs> και του ΕΛΚΑ. Ε, ζητώ συγγνώμη εξ ονόματο της συναδέλφου Ρόζα Εσταράς Σεφεραγκούτ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αιθιοπία με μια ειδική επιστολή και δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα διαβάσω κάποιες ε, παρατηρήσεις τη που μου έδωσε στο γραφείο μου. Σήμερα οι αρχές, οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές έχουν πάνω από 500.000 ε, παράνομους μετανάστες. Περίπου το 40% εξ αυτών ε, παναπατρίζεται στις χώρες προέλευσης ή στις χώρες από τις οποίες ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς την Ένωση. πολιτική, μια αποτελεσματική πολιτική επαναπατρισμού που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα παίζει θεμελιώδη ρόλο για την μεταναστευτική πολιτική που ταυτόχρονα θέλουμε να είναι συνεπής αλλά και ανοιχτή. Στα τέλη του 2010 άρχισαν να ισχύουν οι κοινοί κανόνες ε, περί της επιστροφής ή επαναπατρισμού που έχουν εγκριθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008. Η οδηγία ορίζει κανόνες σαφής διαφανείς και ισορροπημένους όσον αφορά την ε, έκδοση ή την, ε, τον ε, επαναπατρισμό η χρήση καταναγκαστικών μέτρων, ε, η φυλάκιση, ε, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ε, ελευθεριών είναι σημαντικός, κυρίως για τις γυναίκες που είναι πολλές. Θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά μέσω μιας γενικότερης ολοκλήρωσης. Σαν Επιτροπή Γυναικών ε, εγκαλούμε τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές ώστε να λάβουν υπόψη την, τον ευάλωτο χαρακτήρα ε, των ζωών πολλών μεταναστών και θα αναφέρω όλος ιδιαίτερος τις έγκυες γυναίκες και τους ε, ηλικιωμένους που δεν είναι αυτόνομοι και τα θύματα βίας λόγω φύλου θα θέλαμε να η κράτηση των μεταναστών αυτών να είναι η ίστατη λύση και καλούμε τα κρατημέλη να αξιολογήσουν όλες τις πιθανές εναλλακτικέ σε συνεργασία με τις ΜΚΟ του τομέα. Η επαφή με άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όπως οι γυναίκες που είναι σε ενδιαφέρουσα ή που δεν είναι αυτόνομες ή μόνοι γονείς με ανήλικα παιδιά ή ακόμα και και τα θύματα σεξουαλικής βίας ή βίας λογοφύλου σημαίνει την ανάγκη ε, να καταρτιστούν ε, ικανοί υπάλληλοι που να είναι σε θέση ε, συνειδητά να ασκούν τις, τα καθήκοντά τους. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε από την Κομισιόν και τα Κάτι μελη να συνεργαστούν με στόχο να εγγυηθούν μια κατάλληλη κατάρτιση για αυτό το θέμα. και τα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και ε, το θέμα του φύλου. Ε, τέλος, έχουμε αγωνιστεί ώστε οι Κομισιόν από τη μια πλευρά και τα κράτη-μέλη από την άλλη να έχουν υπόψη τους ε, κατά τη διάρκεια της ε, διαβούλευσης για συμφωνίες ε, συνεργασίες με τρίτες χώρες να έχουν υπόψη τους ακριβώς την διάσταση του φύλου. Ευχόμεθα τέλος την εφαρμογή μιας ε, πολιτικής επιστροφής με ανθρώπινο πρόσωπο που να προσαρμοστεί στην ισχύουσα νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ε, ενσωματώνει απολύτως το θέμα, τη διάσταση του φύλου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ματέρα. Και τώρα έχετε το λόγο. Η Κομισιόν έχει να πει κάτι. Έχετε να μας πείτε κάτι, κάποιο σύντομο σχόλιο. Ε, thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σας πω ότι όσον αφορά την οδηγία επιστροφής, συμφωνούμε απόλυτα με τις προτάσεις της Επιτροπής αυτής στο σχέδιο έκθεση, Όντως, η οδηγία επιστροφής έχει τεράστιο δυναμικό προστασίας των ε, παράνομων μεταναστών. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ εκτενές πρόγραμμα εργασίας για την ε, μεταφορά της ε, οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και μπορώ να σας πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στα κράτη-μέλη. Θα παρουσιάσουμε μία έκθεση, μία αίτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και η συνολική μας εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο ε, δυναμικό βελτίωσης, μεγάλες πιθανότητες βελτίωσης. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, όμως μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χρονοδιάγραμμα τώρα, προθεσμία Υποβολή τροπολογιών αύριο 27 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου. Θα ε, ψηφιστεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, την αρμόδια Επιτροπή, στις 16 ε, Ιανουαρίου και δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι πότε θα πάει έκθεση στην Ολομέλεια, να σας πω. Αυτά με το θέμα 14. Προχωράμε στο σημείο 15, συμμετοχή της Ένωσης στην υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση και την έρευνα και ανάπτυξη ε, προγραμμάτων κοινών και από κοινού στα κράτη-μέλη. Κυρία Παλιαδέλη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Λοιπόν, το θέμα μας αφορά την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πρόγραμμα που αναφέρεται στην ε, δραστήρια και υποβοηθούμενη διαβίωση και που επικεντρώνεται όχι μόνο στην έρευνα αλλά και στην εφαρμογή καλών πρακτικών προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα. Είναι μια, Είναι μια γνωμοδότηση που μας ζητήθηκε από την Ήτρε για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πρόγραμμα που έτσι κι αλλιώς διενεργείται από 23 μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το 24ο μέλος αυτής της, ε, ε, αυτού του προγράμματος μετέχοντας ε, στην ουσία ως να ήταν κράτος μέλος προκειμένου να προχωρήσει. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και από τα εθνικά και από τα κράτη-μέλη, από τους μετέχοντες σε εθνικό επίπεδο αλλά και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στον ορίζοντα 2020, στο καινούριο επταετές. Έχει ήδη αξιολογηθεί από μια η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία είδε πολύ καλά πράγματα και συνιστά την ενίσχυση του προγράμματος αυτού, το οποίο στηρίζεται στο ε, άρθρο 185 της Συνθήκης για, την για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της ε, ε, των 28, η συνδρομή θα καταβάλλεται από πιστώσεις του Γενικού Προϋπολογισμού ε, της Ένωσης μέσα από το πρόγραμμα Horizon 2020. Το κείμενο είναι καθαρά ρυθμιστικού χαρακτήρα, επομένως η γνωμοδότηση δεν είχε πάρα πολλές, που και δεν είχε πολλές δυνατότητες για τροπολογίες. Όμως κατατέθηκαν ε, πέντε από τη δική μου μεριά ε, ως εισηγήτριας της νομοδότησης, οι οποίες εστιάζονται σε δύο θέματα. Πρώτον, στη συμμετοχή των γυναικών στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του προγράμματος ε, ζητούμε δηλαδή όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες να μετέχουν και χάραξη πολιτικής και δεύτερον στις υπηρεσίες που παρέχονται στους αποδέκτες όχι μόνο της τρίτης ηλικίας αλλά και του άμεσου περιβάλλοντός τους ε, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία διάκριση για λόγους ηλικίας, φύλου, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικού ή σεξουαλικού προσανατολισμού σε ό,τι αφορά ε, την ε, αποδοχή αυτών των υπηρεσιών. Περιμένω τις δικές σας τροπολογίες, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν νομίζω μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, μέχρι και αύριο δηλαδή, προκειμένου να βελτιώσουμε, αν μπορούμε ακόμα περισσότερο, ένα κείμενο το οποίο δεν μας άφηνε πολλές δυνατότητες παρέμβασης. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Εκπρόσωπω την ε, Γαμαδέλτα Connect, την αρμόδια διεύθυνση. Το πρόγραμμα, με λίγα λόγια, έχει στόχο να καταπολεμήσει τις ε, προκλήσεις ε, της ε, γύρανσης και της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών από τους ηλικιωμένους. Προσπαθούμε να κάνουμε τις υπηρεσίες αυτές πιο ελκυστικές για τους ανθρώπους αυτούς και να λάβουμε υπόψη επίσης και την έμφυλη διάσταση. Επίσης η Γαμαδέλτα μας ασχολείται και με παρεμφερή προγράμματα που αφορούν τις γυναίκες. Τώρα όσον αφορά την δομή της διακυβέρνησης του προγράμματος αυτού, να σας πω ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται στο εκτελεστικό συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης εμείς διασφαλίζουμε ίση εκπροσώπηση στα συμβούλια και στα ε, πάνελ διεξάγουμε αξιολογήσεις τακτικά και εμείς είμαστε εκείνοι που τους διεξάγουμε άμεσα. Όπως σας είπα, στα προγράμματά μας εξετάζουμε το, τη συμπερίληψη των γυναικών και την ίση εκπροσώπησή τους. Επίσης, χρησιμοποιούμε τον ε, κανονισμό για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές που αυτό ορίζει, λαμβάνοντας υπόψη επίσης ε, ζητήματα θρησκευτικού και έμφυλου χαρακτήρα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις ε, τροπολογίες ήδη ε, χρησιμοποιούνται από εμάς, αλλά με χαρά μας να τα επανεξετάσουμε και να τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα ήθελατε να κάνετε κάποια τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, από τη στιγμή που ο στόχος της νομοδότησης ήταν να υποστηρίξει αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολούμαστε εδώ στην Επιτροπή ε, γυναικών. Εκτιμώ ότι η ήδη καλή πρακτική ε, όπως εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια εγγύηση ότι οι τροπολογίες θα γίνουν αποδεκτές και από την Ήτρε και επομένω και από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, προθεσμία υποβολής τροπολογιών αύριο 27 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η Επιτροπή θα ψηφίσει στην επόμενη συνεδρίασή της στις 16 Δεκεμβρίου, η Ήτρα θα ψηφίσει στις 19 Ιανουαρίου και η Ολομέλεια θα ψηφίσει μάλλον το Μάρτιο. Ολοκληρώνουμε με το σημείο 15, περνάμε στο σημείο 16. 7η και 8η έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχή της Ένωσης και στρατηγική, έκθεση στρατηγικής για το 2013 όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων για το 2007 στο 2013. Η κυρία Μπλενκεβίσιουτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ δυνατότητα που μου δώσατε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για το γεγονός πως έχουμε μια τέλεια έκθεση και πλέον πλησιάζουμε και το τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 7-2013 και θα δούμε πώς τα χρηματοδοτικά μέσα ε, συνεισέφεραν στην ε, σύγκληση ε, στις περιοχές αυτές ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης και να δούμε ποια θέματα θα συζητήσουμε πιο πολύ και ποια βρίσκονται στην προτεραιότητα των κρατών μελών. Είπα πως για τα θέματα του φύλου αυτά τα αναφέρονται στις αρχές που διέπουν την ίδια την ύπαρξη των διαστατικών ταμείων. Θεωρούνται ένα αναπόσπαστο σημείο της χάραξης πολιτικής και επαναλαμβάνω εδώ πως παρόλο που οι γυναίκες σε πλειοψηφία έχουν περισσότερα ε, ακαδημαϊκά προσόντα, είναι, πιο, είναι λιγότερο δραστήριες σε επαγγελματικό επίπεδο και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διακρίσεις στις περιοχές της υπαίθρου όπου υπάρχει κίνδυνος πολύ μεγαλύτερος για απόλυτη φτώχεια και πολύ περισσότερες γυναίκες παρά άντρες δουλεύουν σε ε, συνθήκες ε, δύσκολες. Οπότε για το πρόγραμμα 713 η αξιολόγηση που γίνεται αποκαλύπτει πως τα κράτη-μέλη σε γενικές γραμμές κατανόησαν τι σημαίνει ισότητα των φύλων, αλλά και το λέει και η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής είναι ανεπαρκής. Δηλαδή, δεν έχει ενταχθεί αρκετά στα προγράμματα συνοχής η φιλετική διάσταση, η έμφυλη διάσταση. Καλό λοιπόν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες που κάνουν για να κλείσουν το κενό αυτό και να προωθήσουν την οικονομική ε, αυτονομία των γυναικών, να κλείσει λοιπόν το ψηφιακό κενό, το e-gap, και να δούμε και το θέμα της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης και πώς αυτό επηρεάζει τις γυναίκες. Θα ήθελα να καλέσω να καταστήλουν την ε, μεγαλύτερη γυναική αυτόχεια και πιστεύω πως αυτή τη στιγμή η γνωμοδότηση καλεί τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά ταμεία με πιο δραστήριο τρόπο έτσι ώστε να έχουν πολιτικές οι οποίες είναι φιλικές προς την οικογένεια με ε, δομές φροντίδας και μέρημνας για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους και τα υπόλοιπα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Μόνο έτσι θα δώσουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα που είναι ε, πολύ εκπαιδευμένες να συμφιλιώσουν την οικογενειακή και την εργασιακή ζωή και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Και τέλος, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί πιο δραστήρια με τα ευρωπαϊκά όργανα για την ισότητα των φύλων έτσι ώστε να βελτιωθούν τα συστήματα υποβολής εκθέσεων και στοιχείων των ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί ακόμα δυσκολευόμαστε να αξιολογήσουμε την ε, συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Ευχαριστώ και πιστεύω πως πολύ πρόοδο μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα. Και μια τελευταία παρατήρηση, επειδή έχουμε πολύ περιορισμένο πεδίο στην υποβολή τροπολογιών. Κάποια θέματα δεν τα συζήτησα μεν ε, στην, ε, στο κείμενο αυτό. Πάντως θα καλέσω και τους συναδέλφους και τους κοιόδες εισηγητές να το κάνουν έτσι ώστε η δική μας ε, γνωμοδότηση να πάει στην Επιτροπή Περιφερειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί πραγματικά αντιμετώπισε σφαιρικά το θέμα της ισότητας όπως αξίζει και συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία ανέφερε ότι είναι προκλήσεις και πρέπει να τονιστούν στη δική μας νομοδότηση. Εγώ κύριε Πρόεδρε απλά θέλω να τονίσω ότι επειδή η αρχή της ισότητας και η υποστήριξη των δράσεων που αναφέρονται για τη διευκόλυνση της ζωής των γυναικών ή είναι δράσεις που απορρέουν από πρωτοβουλίες των γυναικών είναι αρχές αυτές καταγεγραμμένες στα διαφορετικά ταμεία. Είναι ώρα, την στιγμή αυτή που πάμε σε μια νέα προγραμματική περίοδο, με λιγότερους πόρους, πιο στοχευμένους, με αιρεσιμότητα, ε, είναι ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό της εφαρμογής αυτής της αρχής των διαφορετικών ταμείων στην ισότητα και να εστιαστούμε στις πραγματικές ανάγκες και κενά που είχε αυτή η εφαρμογή. Φυσικά δεν είναι ομοιόμορφα παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά παντού έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες αξιολογήσεις ότι λείπουν τα κατάλληλα εργαλεία από έρευνες, δεδομένα, στατιστικά στοιχεία, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσο τι impact, πόσο ωφελήθηκαν οι γυναίκες από τις δράσεις των διαφορετικών ταμείων πόσο οι δράσει είχαν αποτέλεσμα στη συμφιλίωση τη επαγγελματική και τη οικογενειακή ζωή, πώ αξιοποίησαν το γυναικείο ταλέντο, πώ δημιούργησαν ευκαιρίε για τι γυναίκε επιχειρηματίε. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει πια να τα δούμε με ε, συγκεκριμένα εργαλεία. Είμαστε σε μια περίοδο με τις συνέπειες και τις πληγές της κρίσης ακόμη ζωντανές σε όλες τις περιφέρειες, κυρίως στις περιφέρειες κάποιων χωρών, όπως είναι οι χώρε του Νότου, η χώρα μου ιδιαίτερα, και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πλούτος γυναικείος σε πολλούς τομείς, από την έρευνα, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, κυρίως σε τομείς όπως είναι οι πολιτισμικές και οι δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες είναι, ε, το, βρίσκονται στη, στην περιφέρεια, δίνουν τεράστιες ευκαιρίες για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, συνδυάζονται με τον τουρισμό. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία για να τα αξιοποιήσουν στη νέα προγραμματική περίοδο οι γυναίκες καλύτερα πρέπει πράγματι να δούμε σε αυτό το 7ο και 8ο report ε, τι πρέπει να εντάξουμε σαν κενά και σαν παρακαταθήκη και προτάσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Έχει κάποιος να πει κάτι από την Κομισιόν, παρακαλώ. Γεια σας, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με πολλές από τις ε, ε, αναφορές στην σχέδιο γνωμοδότησης, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ε, το φύλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θέμα οικονομικής προσαρμογής, προκαλώντας έτσι την καταστροφή διαφόρων δυνατοτήτων και δυσχεραίνοντας την αντιμετώπιση προκλήσεων που έχουν αυξηθεί λόγω της κρίσης όπως η φτώχεια. Επίσης συμφωνούμε για τη βελτίωση της παρακολούθησης όσον αφορά την ισότητα των φύλων και ιδιαίτερα έχουμε συμπεριλάβει στην πρότασή μας και για τη μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής συνοχής ένα νέο πλαίσιο απόδοσης που στόχο θα έχει να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματα υπό την πολιτική συνοχή θα αποδίδουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να μετρηθούν αυτό ήταν μεγάλη βελτίωση που καλύπτει το κενό όσον αφορά την ενημέρωση, της προτάσεις ε, με βάση την εμπειρία από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Τώρα εργαζόμαστε λοιπόν με την έκτη έκθεση περί συνοχής, μέτρα που αφορούν το περιφερειακό επίπεδο ΝΑΤΣ 2, ε, και η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο εργάζεται για την διαπραγμάτευση συμφωνιών εταιρικής σχέσης που ξεκινά από την ανάλυση των ε, στόχων ανάπτυξης, των αναγκών μάλλον, των αναπτυξιακών αναγκών και εκεί όπου το θέμα του φίλου είναι ζήτημα, αυτό θα αντανακλάται στα προγράμματα που θα ξεκινήσουν ε, τον επόμενο χρόνο επί τη βάση αυτής της αναλυτικής δουλειάς και των διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. κυρία Βρυνκιβιτσούτη, θέλετε να επανέλθετε και να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ σύντομα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, σκιώδη συγγήτρια, την κυρία Κράτσα, με την οποία συμφωνώ ότι πρέπει να εστιάσουμε στα κενά που υπάρχουν στην εφαρμογή, όπως είπατε κι εσείς, διότι ε, μόνο εάν όντως αντιμετωπίσουμε αυτά τα κενά, τα κενά μπορούμε να αποφύγουμε τα ίδια λάθη στη νέα προγραμματική περίοδο. Πιστεύω πως ε, συνεργαζόμενες θα μπορέσουμε να φτιάξουμε συμβιβαστικές προτάσεις για το κείμενο αυτό και ευχαριστώ και την Κομισιόν διότι συμφωνώ μαζί σας ότι τα προγράμματα θα πρέπει εξ αρχής να ε, περιλαμβάνουν κάποιους δείκτες, να ορίζουν κάποιους δείκτες, ώστε να μπορούν αυτοί μετά να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του προγράμματος, το οποίο έχει λάβει κάποια χρηματοδότηση. Να δούμε κατά πόσο έχει πετύχει τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, χρονοδιάγραμμα Σαν παπαγάλος ακούγομαι γιατί όλα τα ίδια λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι η τελική προθεσμή για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο 27 ε, Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, θα ψηφίσουμε στις 16 Δεκεμβρίου και η Ρέτζη θα ψηφίσει 22 και 23 Ιανουαρίου και θα περάσει από την Ορλομέλεια από όσο ε, φαίνεται τον Φεβρουάριο. Έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε και το 17 που αφορά την επόμενη συνεδρίαση με κοινή συνεδρίαση ανάμεσα στην Επιτροπή μας και την Επιτροπή Αλληλείας. Για αύριο από τις 10 με... Ε, μέχρι 11 και 50, ε, συγγνώμη 10 και 50 και Έχουμε και άλλες συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου στις 5 Δεκεμβρίου αλλά και στις 16 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ, καλή σας όρεξη.